Βέβαια έχουμε μια, μεγάλο, μια μεγάλη ποσότητα η οποία οδηγείται στην κονσερβοποιία. Είναι ε, η, εκτροφή του, του τόνου είναι αυτή η οποία έχει την μεγαλύτερη εμπορική αξία και έχουμε 65.000 τόνου τόνους ετησίως. Αυτή τη στιγμή η ICAT ελέγχει την, ε, την, τα, και την εκτροφή αυτών των ειδών. Ε, έχουμε πολύ αυστηρούς ελέγχους που και υπάρχει και ένα σχέδιο για την αύξηση των ποσοτήτων. Για την αύξηση των αποθεμάτων τώρα για, την, για τον ερυθρό τόνο του, του ειρηνικού δεν υπάρχει κανένα σύστημα ποσοστώσεων που να έχει εφαρμοστεί. Ε, τα αιτήσια αλλιεύματα είναι περίπου 20.000 τόνους. Αυτή τη στιγμή ε, για τον ε, Ανατολικό Ατλαντικό και τα αποθέματα ε, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ότι είχε καταλήξει στο ΙΑΙ e κάτω το 2010 στην ε, μελέτη που είχε κάνει. Για τα αλλιεύματα είναι λιγότερο από 12.000 τόνους ε, μέσα στα πλαίσια δηλαδή των επιστημονικών συμβουλών. 180.000 τόνοι για την βιομάζα ανα αναπαραγωγής ε, έχουν υπολογιστεί για το 2010 από την ΆΕΚΑΤ, δηλαδή ε, αυξήθηκε, διπλασιάστηκε από, τα τελευταία, από την τελευταία ε, χρονιά αναφοράς η προηγούμενη εκτίμηση που είχε γίνει το 2008 με τα πραγματικά στοιχεία που είχαμε μέχρι το 2006 ε, ανήρχεται σε 78.000 τόνους. Τώρα, όσον αφορά τα αλλιεύματα, βρισκόμαστε σε ιστορικά χαμηλά νούμερα, ε, ούτε τη δεκαετία του 70 δεν τα είχαμε αυτά, ε, διότι υπάρχει ένα σύστημα, ε, ναι, ένα, σύστημα αναγέννησης των αποθεμάτων ε, και ελπίζουμε ότι τα, τα αποθέματα θα έχουν ε, φτάσει στα όρια τα οποία θέλουμε μέχρι το 2022 έτσι ώστε να έχουμε μια μέγιστη απόδοση 50.000 τόνων από το 2023 και μετά. Τώρα όσον αφορά την εμπορική ε, τις εμπορικές κατηγορίες έχουμε τον κονσερβοποιημένο τόνο, την αγορά για τις ε, κονσέρβες που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι μετά έχουμε ε, την αγορά για, την, για τα φιλέτα τόνου και μετά έχουμε και την αγορά για τον ομό τόνο ο πιο ακριβώς είναι ο ερυθρός τόνος βλέπετε στην ιαπωνική αγορά μετά έχουμε τον νότιο τόνο, ε, ο μεγαλόφθαλμος ε, επίσης ακολουθεί και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει και το πιο ακριβό είναι, το, είναι ο τόνος ο οποίος προορίζεται για τα σούσι και τα σασίμι. 20, ευρώ το κιλό είναι η τιμή λίγο πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, προφανώς, ε, η, ο τόνος για το σούσι και το σασίμι στην Ευρώπη ε, δεν, ζητά, δεν ζητείται πολύ και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουμε λίγο πολύ 4.000 τόνους για το τόνο για το σασίμι. Όπως σας είπα, 20.000 τόνοι είχαν αλλιευθεί πέρυσι. 30 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτό, μέσα στα πλαίσια αυτού του αποθέματος έχουμε ε, και τις δραστηριότητες πάχυνσης. Επίσης αυξάσαμε την τιμή από 6 ευρώ σε 20 ευρώ και αυτό γιατί διότι όσον αφορά τα άγρια αλλιεύματα, μονάχα ένα κομμάτι, ένα τμήμα προορίζεται για σούσι και σασίμι, λόγω ακριβώς των συνθήκων που επικρατούν πάνω στο πλοίο. Επίσης, αυξήθηκε και το ποσοστό λίπους. Έχουμε μια μεγάλη προστιθέμενη αξία, αν θέλετε, πολύ περισσότερη από οποιαδήποτε άλλο, άλλη δραστηριότητα που αφορά τον τόνο και την, ε, και την εκτροφή του. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο τομέας αναγκάστηκε να περιορίσει τον όγκο των αλλιευμάτων και υπήρξαν, ε, υπήρξε μια αναδιάρθρωση του τομέα. Ε, η παραγωγή και οι πωλήσει περιορίστηκαν πάνω από 50% το 2010 σε σχέση με το 2006 είχαμε σημαντικές μειώσεις ε, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι ο τομέας αυτός ε, θα το από αυτή την αύξηση των τιμών ε, και με την περιορισμένη, λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη ε, προμήθεια στην αγορά. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν, σημαίνει, δεν συνέβη διότι οι, οι ανταγωνιστές στο τομέα εκτροφής του τόνου με την βοήθεια κιόλας των κανονιστικών ελλημάτων που είχαμε στον, στον ειρηνικό αύξησαν σημαντικά την παραγωγή τους και κάλυψαν το κενό. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών και το κόστος των νέων μέτρων και οι διαδικασίες που επιβλήθηκαν ε, καταλήξαμε σε κάποιες οικονομίες κλίμακας οι οποίες επιδίνωσαν και ε, περιόρισαν τα περιθώρια κέρδους. Επίσης ε, ε, η, η, εκστρατεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, ανάγκασε την ευρωπαϊκή και μεσογειακή βιομηχανία να περιορίσει σημαντικά τους όγκους της τα τελευταία χρόνια και αυτή η εκστρατεία έδειξε ότι ήταν επιλεκτική και επέβαλε διακριτική μεταχείριση. Σας είπαμε ότι ήταν ε, η εκστρατεία αυτή ήταν αρνητικά, είχε αρνητικές συνέπειες και το μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Ήταν προκατηλημένη και το, τα αποθέματα το 2009 περιορίστηκαν ε, στο 20% των ε, ιστορικών ορίων Τώρα όμως βλέπουμε ότι έχουμε μία αύξηση που, φτάνουμε στο 57, που έχουμε φτάσει στο 57% και το επίπεδο αυτό αυξάνεται. Πιστεύουμε ότι, τα... ότι θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση αν είχαμε, στη συγκεκρι... είχαμε τη συγκεκριμένη στιγμή της λήψης των αποφάσεων είχαμε τα πραγματικά στοιχεία. δεν, ε, ε, δεν ζητήθηκε ένας κατάλογος για να έχουμε τα στοιχεία που αφορούν ε, τον ερυθροτόνο και θα θυμόσαστε ότι, το 2000, ότι το, η Σουηδία είχε ζητήσει να καλυφθούν όλες, όλες οι κατηγορίες. Επομένως, γιατί δεν πήραμε τα στοιχεία από τόνους και επικεντρώσαμε την προσοχή μας μόνο στον ευρωπαϊκό μεσογειακό τόνο, ε, τώρα, το πρόβλημα είναι πώς ε, μπορούμε εμείς να απαντήσουμε. Ε, μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έγινε ήταν να αποκρυβούν κάποια, κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε στις 11 ε, Νοεμβρίου του 2010 πριν από την ετήσια σύνοδο της ΆΕΚΑΤΑ το Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ε, την ε, απογραφή που έγινε στο τέλος του Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς οδήγησαν σε αυτή εδώ την γραφική παράσταση που βλέπετε εδώ ότι σα είπαν δηλαδή τότε ε, ότι η κατάσταση είναι δραματική, όμως σα απέκρυψαν το γεγονός ότι, είχαμε φτάσει, ότι το, τα αποθέματα δεν ε, αντιμετώπιζαν οποιοδήποτε κίνδυνο εξαφάνισης. στη γραφική παράσταση που βλέπετε τώρα, βλέπετε τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει στην ΆΕΚΑΤ όταν προσπάθησαν να αναλύσουν τα στοιχεία της αγοράς που προέρχονταν από την Ιαπωνία ε, για τον ε, ερυθρό τόνο και έδειξαν εκεί ότι τα αποθέματα αυτά μειώνονται. Βλέπετε τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα, τα οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ε, γιατί έχουμε μονάχα ένα εκτροφείο, το οποίο εγώ διαχειρίζομαι ε, λέγεται ότι από το 2008 έως το 2009 ε, εξάγαμε 4.000 τόνους. Αυτό, αυτή είναι η πληροφορία που έδωσαν στον ΆΙΚΑΤΑ. Όμως όλα αυτά τα στοιχεία για τα ψάρια τα οποία έδειξαν ότι 66 κομμάτια, πολλά από αυτά μικρού μεγέθους, Πόσα όμως ε, εξήγαμε στην Ιαπωνία στο δεύτερο ήμιση του 2008, εμείς μηδέν. Και όμως ε, έδωσαν αυτές τις προφορίες στον ΆΕΚΑΤ και στο πρώτο εξάμεινο του 2009 για να σας δείξω δηλαδή την ποιότητα των στοιχείων που δείχνουν, ε, που έδωσαν αναφέρονται κάποιες εξαγωγές ε, οι οποίες αποκλίνουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. Δηλαδή μας είπαν ότι εμείς ε, ε, εξήγαμε 66 ζώα τα οποία δεν, δεν εξήγαμε κανένα, ενώ το, τη δεύτερη χρονιά μονάχα το, αναφέρουν ένα ποσό που αφορά μονάχα το 10% των όσων έχουμε αλλιεύσει. Τώρα, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τον, τον ερυθρό τόνο, Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η, από την αρχή της δεκαετίας του 70 το, τα αποθέματα για τον ερυθρό τόνο έχουν περιοριστεί κατά 80% ενώ κατ' ουσίαν έχουν περιοριστεί μόνο κατά 43%. Επίσης για τα λιεύματα να φέρουν ένα ποσοστό 70% ενώ είναι μόνο 50% βλέπετε την μείωση στην συνολική παραγωγή εκτρεφωμένου ερυθρού τόνου και βλέπετε για την Ιαπωνία λόγω ακριβώς των κανονιστικών ρυθμίσεων και λόγω των ε, στοιχείων που έδωσαν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και που αφορούσαν τον ευρωπαϊκό και μεσογειακό τόνο. Είχαμε διάφορε αρνητικέ ε, συνέπειε. Βλέπετε η Ισπανία, η Μάλτα και η Κροατία και μετά είναι η Τουρκία είναι οι μεγαλύτερε ευρωπαϊκέ χώρε παραγωγή. Όπως ε, Αναφέρονται, αναφέρεται και από την Επιστημονική Επιτροπή της ΆΙΚΑΤ ο, ο ανατολικός άγριος τόνος και τα αποθέματα του ε, μειώνονται αλλά δεν, ε, αυξάνονται και δεν, έχουν, δεν ε, ε, αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε κίνδυνο κατάρρευσης ε, σύμφωνα με, με το τρέχον ΤΑΚ και τα μέτρα ελέγχου και συμμόρφωσης που έχουν εφαρμοστεί. Η Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να ε, θεωρεί ότι θα έχουν ε, ε, δημιουργηθεί ξανά τα αποθέματα μέχρι το 2022 σε ένα μέγιστο επίπεδο βιωσιμότητας με απόδοση 50.000 5.000 τόνους από το 2023 και μετά ε, η παραγωγή και εκτροφής ευρωπαϊκού τόνου θεωρούν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις αρχές της βιωσιμότητας και της συχνηλεσιμότητας ε, μέσα στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης ε, εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αγρίου τόνου και ζητούν προφανώς την υποστήριξη της Επιτροπής Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε σε δύο-τρία χρόνια να μην εξαρτώμεθα από, την, από τον άγριο τόνο. Και να σας δείξω και ποιες είναι οι δραστηριότητές μας. Βλέπετε, μια, βλέπετε την, ένα τόνο, βλέπετε τα, τα λιευτικά σκάφη, βλέπετε τα γρηγρή πώς αλλιεύουν, βλέπουμε την, τον τρόπο με τον οποίο τα κλουβιά τα, έχουν, είναι κατεστημένα, πώς γίνεται η τα κτλ. Βλέπετε εδώ μια, ένα εκτροφείο, κλασικό εκτροφείο, απλώς εδώ τα κλουβιά είναι πολύ μεγαλύτερα λόγω του ότι είναι μεγαλύτερο και το ζώο. Βλέπετε τις δραστηριότητες εκτροφής, πώς τα, τα ταΐζουν τα, τα ζώα. Βλέπετε πώς αλλιεύονται τα, τα ψάρια τα οποία αλλιεύονται και, τα, και παραδίδονται σε αλλιευτικά ιαπωνικά σκάφη, ψυγεία, τα οποία καταψύχουν αμέσως τον τόνο στους μείον 60 βαθμούς. Ε, η, η παραγωγή ε, τόνου, μάλλον η πώληση τόνου ε, γίνεται αυτή τη στιγμή σε υπομορφή κατεψυγμένου προϊόντος στους μείον 60 βαθμούς και μπορεί να παραμείνει το ζώο για 2-3 χρόνια στην ε, κατάσταση αυτή ενώ εάν είχαμε μείον 18 βαθμούς σε ένα μήνα περίπου το προϊόν θα καταστρέφεται. Και ήθελα να σας πω ότι εμείς κρατάμε το ζώο για ένα χρόνο και μας παρακολουθούσαν ε, οι παρατηρητές, ε, γίνανε ντοκιμοντέρ, ε, γυρίστηκαν ταινίες και όλα αυτά με υψηλό κόστος. Οι Ιάπωνες εμποροί, οι Ιάπωνοι κρατάνε το προϊόν για στους μείον 60 βαθμούς για τρία χρόνια και εκεί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ε, δεν ελέγχονται από την ΆΙΚΑ τα ψυγεία, δεν υπάρχουν παρατηρητές, δεν ελέγχουν τα, τα έγγραφα κτλ. Αυτό το έχουμε πει στην Κομισιό, αλλά δεν ε, μπορούν να επιβάλλουν ελέγχους προφανώς στην, στα ιαπωνικά ψυγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Περνάμε στον επόμενο που είναι ο κύριος Χουάν Σεράνο Φερνάντες, πρόεδρος της ομάδας Μπαλφεγό. Έχετε το λόγο λοιπόν για 10 λεπτά περίπου. Παρακαλώ. Ya está, Señora Presidenta, señoras y señores diputados. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες βουλευτές, εποφελούμαστε από την ευκαιρία αυτή για να σας παρουσιάσουμε κάποια θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση της Αγγλίας γενικότερα και πιο συγκεκριμένα του ερυθρού τόνου. Η ομάδα μου είναι η πέμπτη γενιά αλλιών που ξεκίνησε τη δραστηριότητά τους πριν από 15 χρόνια στη Μάγια Δεμάρ, στην Ταραγώνα. Και χάρη στις προσπάθειές μας, ε, στη, στο επιστημονικό μας ε, όραμα και στη βοήθεια που είχαμε, από το 2004 έχουμε δύο αλλιευτικά σκάφη ένα, και μια επιχείρηση, μια ελευτική και σιγά σιγά θα πάρουμε και άλλα δύο σκάφη. Η πρώτη αλής ξεκίνησαν με την αλλαγή στην κατάσταση του ερυθρού τόνου στην Μεσόγειο. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από την αλίευση και φτάνουμε στον τελικό καταναλωτή για τον ερυθρό τόνο. Αλλά συγχρόνως ήμασταν οι πρώτοι που προτείναμε μέτρα διαχείρισης και ελέγχου για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός από αυτούς που δεν τηρούν τους κανόνες. Μέτρα λοιπόν τα οποία ως επιτοπλίστων ισχύουν σήμερα. Πρώτα απ' όλα ε, ηλεκτρονικά να μπορεί να ελέγχεται ο τόνος σε όλες τις περιοχές όπου αλλιεύονται μέχρι που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή με διαφάνεια. Έτσι η πληροφορία αυτή υπάρχει και στη διάθεση και των καταναλωτών και όσων διαχειρίζονται τα αλλιευτικά αποθέματα. Και αυτό ακόμα και μέσω κινητού. Παρακολουθούμε την αλίευση σε όλα τα στάδια. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επενδύουν στην αλίευση του ερυθρού οπότε και αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμε. Από 26 που είχαμε στην αρχή έχουμε 200 υπαλλήλου σήμερα σε μόνιμη βάση. Έχουμε την εμπορική μας δραστηριότητα διαφοροποίηση και γεωγραφικά έχουμε διαφοροποιηθεί και είμαστε εκείνοι που εξαρτώμεθα λιγότερο από την Ιαπωνική αγορά. 44% της παραγωγής μας και 22% είναι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εμείς καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς. Εισάγουμε ε, εισαγόμαστε μάλλον σιγά σιγά ακόμα και στην Ιαπωνική αγορά. Τροφοδοτούμε ε, πολλά εστιατόρια σε ολόκληρη την Ευρώπη με προϊόντα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας υπεύθυνα πάντα. Σήμερα εκπροσωπούμε το 18% σε όγκο της ισπανικής ποσόστοσης, πάνω από 50% της αξίας του τόνου που εμπορεύεται η Ισπανία και στην Μάγια Ντεμάρ η δραστηριότητα αυτή έχει τεράστια σημασία για τον τόπιο πληθυσμό. Είμαστε το 20% της καταλανικής αγοράς. Αντιλαμβανόμαστε όμως συγχρόνω ότι ο άνθρωπος προσπαθώντας να πετύχει όλο και περισσότερη ευημαρία πολλέ φορέ καταστρέφει τον ίδιο το χώρο στον οποίο ζει. Οι διερμηνείς δεν σα προλαβαίνουν, λέει η Πρόεδρος. Πιο αργά παρακαλώ. Μα μου είπατε 10 λεπτά. Ε, ναι, αλλά τι να κάνουμε. Ζητάει συγγνώμη ο μιλητή. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε υπεύθυνα να συνεισφέρουμε ώστε το περιβάλλον να το προστατεύουμε και να μην το καταστρέφουμε. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2371 ε, καθορίζει ως στόχο ότι η κοινή ελευτική πολιτική διασφαλίζει εκμετάλλευση των ε, αλληλευτικών πόρων υποστηρίζοντας ε, την οικονομική βιωσιμότητα αλλά προστατεύοντας πάντα το περιβάλλον. Αυτό ακριβώς κάνει η ομάδα μας. Και το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε βασικές αρχές. Μεταξύ άλλων, ακολουθούμε αξίες που είναι η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η υπευθυνότητα. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, γιατί οι πόροι που χρησιμοποιούμε πρέπει να βελτιώνονται, γιατί έτσι διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε επίσης να φροντίζουμε τη σημερινή στιγμή όπου πολλές χώρες όπως και η δικιά μας ε, χάνει ανταγωνιστικότητα εμείς να αυξήσουμε ε, τους πόρους μας. Χωρίς καμιά αμφιβολία, η ελιευτική δραστηριότητα πρέπει να βασίζεται σε οικονομικές ε, λογικές αρχές. Όλοι πρέπει να ενισχύονται οικονομικά, αλλά συγχρόνως να λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον, αλλά και τις αλλαγές των αγορών. Θέλουμε επίσης διαφάνεια, διότι ο καταναλωτής και η κοινωνία πρέπει να έχει ενημέρωση όσον αφορά τις δραστηριότητές μας και δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες μας και στην κοινωνία γενικότερα να καλύπτουμε τις προσδοκίε τους για αηφόρα δραστηριότητα, για βιώσιμη ελεία. Το κάνουμε αυτό στη Μεσόγειο και θέλουμε και υπευθυνότητα γιατί φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες κατά γράμμα και τους νόμους. Θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι γιατί όλους μας όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε τις δραστηριότητε μας με άξονα τη βιωσιμότητα. Η αλία εποφελείται από ελεύθερη πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, αντίθετα με άλλους κλάδους. Συγχρόνως όμως υπάρχει ο έλεγχος στη θάλασσα, που είναι πολύ σημαντικός. Και έπειτα υπάρχουν και επιδοτήσεις στον τομέα. Πάντως, αυτά τα οποία βοηθούν τη βιωσιμότητα του κλάδου είναι τα εξής είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία ε, λαμβάνει χώρα στη θάλασσα. Από τον ε, κανονισμό αυτό λοιπόν, στο τρίτο άρθρο, αναφέρεται η βιώσιμη αλία έτσι ώστε να μην ε, πλήτεται η μελλοντική εκμετάλλευση των πόρων αυτών και χωρίς να καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον. Ο ορισμός της ε, βιώσιμη εκμετάλλευση ή τη βιώσιμη αλίας είναι ένα ορισμό που πρέπει να διαβρεθεί περισσότερο. Γιατί για μα σημαίνει κάθε αλληλευτική δραστηριότητα και εμπορία τη αλληλευτική παραγωγή που επιτρέπει ε, αναζωγόνηση των πόρων, αναγέννηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι αυτοί και για τι επόμενε γενιέ. Και αυτό σημαίνει ότι εμεί πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε και αξία για την κοινωνία και απασχόληση ποιότητας και νέες ευκαιρίες για όλους, προστατεύοντας συγχρόνως τους αλληλευτικούς πόρους. Έτσι λοιπόν, εμείς εμπορευόμαστε τον ερυθρό τόνο υπεύθυνα, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πελατών μας σε συνεχή βάση και διασφαλίζουμε και τη συνέχιση του είδους για να υποφελουθούν από αυτήν οι επόμενες γενιές. Εμείς αλλιεύουμε τόνο χωρίς όμως να ε, πετάμε τόνο στη θάλασσα στη συνέχεια. Προστατεύουμε την ελία αυτή και φροντίζουμε να καταναλώνεται και άμεσα. Σίγουρα είναι ο καλύτερο τρόπο αλία αυτό που χρησιμοποιούμε για τον τόνο, γιατί χρησιμοποιεί και λιγότερα καύσιμα. Τα πληρώματά μα επίση συμμετέχουν στα κέρδη από την αλληλευτική δραστηριότητα. Είναι η δραστηριότητα η οποία προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και μάλιστα ολόκληρο το χρόνο. Είναι οικονομική δραστηριότητα η οποία μας επιτρέπει να βάζουμε σε μια ισορροπία τη ζήτηση και την προσφορά στην απασχόληση. Είναι η δραστηριότητα η οποία δίνει η περισσότερη προσθεθέμενη αξία στην αλία. Η δραστηριότητά μας δεν καταστρέφει πόρους. Αυτός που καταστρέφει πόρους είναι αυτός που είναι ανεύθυνος και σε αυτόν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις και θα πρέπει να εκδιωχθεί μάλιστα και από τη δραστηριότητα. Όσον αφορά τώρα την έρευνα, εμεί πιστεύουμε ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική μια ε, δραστηριότητα, πρέπει να φροντίζει να υπάρχει και έρευνα. Ο Αλιέ δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα στη θάλασσα χωρί να ξέρει πώ πάνε οι πόροι. Πρέπει να ξέρει ποια είναι η εξέλιξη των πόρων. Πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και να συνεργάζεται με του επιστήμονε. Εμεί λοιπόν έχουμε επενδύσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 2 εκατομμύρια και έχουμε φροντίσει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ανανεώνουμε και τον τρόπο διαχείρισης ε, στον κλάδο. Έχουμε 10 επιστημονικά προγράμματα, συνεργαζόμαστε δηλαδή με την επιστημονική κοινότητα για 10 επιστημονικά προγράμματα και με την ΙΚΑ. Μόνο γνωρίζοντας, ε, έχοντας καλύτερη επιστημονική γνώση για την Ελία, μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείρισή της και να πετύχουμε βιωσιμότητα στην Ελία. Και συγχρόνως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κάθε αλίας πόσο μεγάλη σημασία έχει να χρησιμοποιεί σωστά κριτήρια στη διαχείριση ε, της δραστηριότητάς του. Το 2007 ξεκίνησε ένα σχέδιο ανάκαμψης από το οποίο επεφελούμαστε σήμερα. Γιατί αυτό που είναι το πρόβλημα είναι η υπεραλίευση, την οποία την έχουμε ακούσει περισσότερο για τον τόνο. Υπάρχει όμως η αδήλωτη, η μη ρυθμισμένη αλία για πολύ μεγαλύτερη γκάμα ειδών και όχι μόνο για τον τόνο, τον οποίο καταδεικνύουμε συνέχεια. Δεν πρέπει να θεωρείται μόνο δικός μας ο κλάδος υπεύθυνο για την υπεραλίευση, γιατί δεν είναι έτσι. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανεύθυνο. Δεν είναι δυνατόν να δαιμονοποιούμε ε, μία μόνο περίπτωση επειδή ένα μονοκλάδο, επειδή συμβαίνουν ε, καταχρήσεις αλλού. Οι πολιτικές ε, κατά της υπεραλίευσης πρέπει να προχωρήσουν με μέτρα ελέγχου πάνω απ' όλα. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη από 146 πέρασε σε 28 σκάφη και έτσι έχουμε καταλήξει να μειώνουμε και τα λιεύματα. Με τα μέτρα ελέγχου του κανονισμού του 2009 έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Έχουμε την πιο ρυθμισμένη αλία και την περισσότερο ελεγχόμενη στον κόσμο. Τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί περιορίζουν τα λιεύματα και πιστεύουμε ότι είναι ορθά τα μέτρα αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια που δεν εφαρμόζονται αδιακρίτως. Πρέπει να ισχύσει το κριτήριο που μιλάει για την παραμονή στη θάλασσα των σκαφών εκείνων που τηρούν τα κριτήρια για την αηφόρο αλία, τη βιώσιμη αλία και που ακολουθούν τους ίδιους στόχους όπως και το δεύτερο άρθρο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την διατήρηση των ειδών και την ε, αηφόρο εκμετάλλευση των πόρων. Η παράνομη και αδήλωτη αλία πρέπει να καταργηθεί μέσω του κανονισμού του 2009. Να σταματήσει η παράνομη και αδήλωτη και μη ρυθμισμένη αλία. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει συνείδηση σε όλους, από τον αλία μέχρι τον καταναλωτή. Για να σταματήσει η παράνομη αλία Μάλλον για να υπάρχει παράνομη αλεία, υπάρχει κάποιος παράνομος αλείας, υπάρχει κάποιος ε, παράνομος ε, μεταφορέας, αλλά υπάρχει και ένας ασυνείδητος καταναλωτής ή ένας μη καλά πληροφορημένος, ενημερωμένος ε, καταναλωτής. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Για να υπάρχει παράνομη αλεία, υπάρχει κάπου συνενοχή. Εμείς γι' αυτό θέλουμε ελέγχους στα σκάφη μας, στα λιμάνια μας, από την αρχή της δραστηριότητας μέχρι το τέλος, μέχρι το σημείο πώλησης, μέχρι τις αγορές. Η πιστοποίηση που λέει ότι το κάθε προϊόν προέρχεται από βιώσιμη αλεία είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί μια μεγάλη πρόοδο. Ο έλεγχος βέβαια σημαίνει παραπάνω έξοδα. Και παρόλα αυτά δεν φτάνουν. Ενώ στην εσωτερική αγορά, αυτό συμβαίνει στην εξωτερική αγορά για ό,τι βγαίνει, αλλά στην εσωτερική αγορά δεν υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι. Παρ' όλα αυτά, με ελάχιστο κόστος από την κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει αυτό και θα μπορούσε να υπάρχει διαφάνεια στον τομέα. Η ομάδα μας έχει ήδη αποδείξει ότι γίνεται αυτό. Είναι εφικτό στην πράξη. Επιπλέον, έτσι θα βοηθούσαμε και οικονομικά τις κυβερνήσεις. Πριν από λίγο καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε η κυρία Δαμανάκη ότι αυτή η παράνομη αλία θα μπορούσε να μας δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ αν ελεγχότανε. Οι κανόνες πρέπει να φροντίσουν να στηριχθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις, εκείνες που τηρούν τους κανόνες και στην ε, αλήψη και στην μεταποίηση. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ένα αλληλευτικό τομέα απλώς και μόνο με μικρά σκάφη και να προσπαθούμε αυτά τα μικρά σκάφη να τα κάνουμε να τηρούν τους κανόνες ενώ αφήνουμε τα μεγάλα να παρανομούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική σωστή αλία. Ζητάμε δικαιοσύνη για όλα τα σκάφη, για όλους τους τρόπους αλίας πρέπει να υπάρχει μια συγκρίσιμη κατάσταση μεταξύ άλλων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας έναν ε, καλύτερο κόσμο. Αλλά πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε πράξεις ε, ανεύθυνες ή υπεύθυνε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, επιλέγουμε την υπευθυνότητα, την ε, σωστή απόδοση, την ποιότητα. Και ελπίζουμε ότι όλα αυτά που βρίσκονται στα κείμενα θα υπάρχουν και στο πνεύμα της εφαρμογής της, ε, του κάθε κανονισμού και της κάθε ρύθμισης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεράνο. Μας δώσατε το παράδειγμα μιας επιχείρησης όπως είναι η δικιά σας και μας εξηγήσατε τις προσπάθειες που κάνετε για την βιωσιμότητα του κλάδου. Πολύ ενδιαφέροντα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ε, δόκτωρα Άννα Κορδό, που είναι από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους σας. Θα προσπαθήσω σε λίγα λεπτά να σας εξηγήσω τι κάνουμε εμείς στο Μπαλφεγό. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την Παλφεγό από το 2008. Στόχος μας ήταν κάτι πολύ απλό. Ήταν να καθορίσουμε κατά πόσο στους κλοβούς όπου μεταφέρονται τα ψάρια ε, γίνεται και αναπαραγωγή του είδους. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια δειγματοληπτική μέθοδο η οποία θεωρείται επιτυχής. Μας εξέπληξαν μάλιστα τα αποτελέσματα τα οποία ήταν πολύ καλύτερα από αυτά που περιμέναμε εμείς ήδη. Για πρώτη φορά διαπιστώσαμε πώς γίνεται η αναπαραγωγή του ερυθρού και την παρατηρούμε μέσα σε τέτοιους κλοβούς. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι παρατηρούμε ότι γίνεται σε τακτικούς ρυθμούς καθημερινά και έτσι μπορέσαμε να καθορίσουμε ακριβώς πότε αναπαράγεται ο ρυθρός τόνος. Ξεκινήσαμε έτσι μια νέα έρευνα και χρησιμοποίησαμε τους κλωβούς αυτούς σαν βάση για την έρευνά μας. Δεν βλέπετε ολόκληρη τη διαφάνεια, λέει ο Μιλήτρια. Ε, Καλά, θα σας τα πω τότε, αφού δεν τα βλέπετε. Σας είπα ότι τους κλωβούς αυτούς τους χρησιμοποιούμε σαν βάση για την έρευνά μας. Υπάρχουν δύο ειδών έρευνες. Η μία είναι η βασική έρευνα και η άλλη είναι εφαρμοσμένη που κάνουμε με την ομάδα Παλφεγό. Στη βασική έρευνα, πρώτος στόχος είναι να δούμε με ποιο τρόπο γίνεται η αναπαραγωγή του τόνου στις νήσους Βαλεαρίδες. και βλέπουμε πώς και πού είναι ε, παρόντες οι τόνοι. Είναι ένα μεταναστευτικό είδος που πηγαίνει στις περιοχές αναπαραγωγής, αλλά δεν φτάνουν όλοι συγχρόνως. Και εμείς θέλουμε να διαπιστώσουμε ποια στιγμή στις βαλερίδες νήσους υπάρχει η μέγιστη παρουσία αναπαραγωγής, δηλαδή των τόνων που αναπαράγονται. Διεξάγεται η έρευνά μας ε, και με τα αυγά και τους γόνους ε, του τόνου και παίρνουμε δείγματα στη Μεσόγειο για να δούμε αν υπάρχουν γενετικά διαφοροποιημένοι οργανισμοί. Και βλέπουμε πώς γίνεται και η εκτροφή στους κλοβούς. Έχουμε λοιπόν αποτελέσματα από αυτήν την βασική έρευνα και βάσει αυτής βλέπουμε τι αλλαγές υπάρχουν. Θα προσπαθήσω τώρα να σας εξηγήσω αυτή τη διαφάνεια, πώς γίνεται δηλαδή η αναπαραγωγή και η αναδιάταξη. Κάθε χρόνο παίρνουμε δείγματα για το σκοπό αυτό και χρησιμοποιούμε τους κλοβούς τόνων γι' αυτό. Τα στοιχεία που ελέγχουμε είναι οι άγριοι τόνοι που έχουν συλληφθεί πρόσφατα. Οι πρώτοι δηλαδή που φτάνουν στην αναπαραγωγική περιοχή και τους πιάνουμε, μπαίνουν σε κλοβούς και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε τη συμπεριφορά τους μέχρι να ξέρουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή αυτής της ομάδας. Συγχρόνως ελέγχουμε και άλλη ομάδα η οποία ε, πιάστηκε το 2008 και έχει μεταφερθεί μέχρι την ζώνη αναπαραγωγής για να αναλύσουμε και το δικό της τρόπο αναπαραγωγής και να δούμε ποια είναι η εξέλιξη ανάλογα με το πόσο καιρό βρίσκεται στους κλοβούς. Η περίοδος ε, δειγματοληψίας είναι από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μέσα Μαΐου είναι η στιγμή που πιάνουμε τα πρώτα ζώα προς αναπαραγωγή και τον Ιούλιο είναι η στιγμή που εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή αυτής της ομάδας. Όπως σας είπα, η αναπαραγωγή γίνεται καθημερινά και αυτό το διαπιστώνουμε από το 2008. Εδώ έχετε κάποιες εικόνες για να δείτε τους ε, Βλέπετε εδώ τους κλωβούς, τη μεταφορά. Οι διαστάσεις είναι 50 μέτρα ε, διάμετρος. Έχουμε χίλιους τέτοιους κλωβούς. Χίλια, ούτε 10 ούτε 20 κομμάτια. Την νύχτα δουλεύουμε. Εδώ βλέπετε δίκτυα. Βλέπετε ότι είναι στην επιφάνεια για να μπορέσουμε να πάρουμε δείγματα πλακτού όπου βρίσκουμε και τα ΟΑ. Εδώ δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά πρόκειται για ΟΑ, στα οποία, τα οποία τα μαζεύουμε, τους μπαίνουν ετικέτες και πάνε στο εργαστήριο. Αυτά που βλέπετε εδώ το λευκό είναι αυγά. Γίνεται έρευνα ε, τόσο στα εργαστήρια, στη Ξηρά, αλλά και στα σκάφη μας ε, στη θάλασσα. Στο Ισπανικό Κέντρο Κενογραφίας, για παράδειγμα, γίνονται έρευνες. Τα μαύρα κομματάκια που βλέπετε είναι γόνοι. Εδώ βλέπετε το περιεχόμενο του στομαχιού. Υπάρχει πολύ πλαστικό μέσα, όπως ε, βλέπετε. Και κάτι άλλο που βλέπουμε σε αυτή την περιοχή συστηματικά και όλο και περισσότερο είναι μέδουσες. Διαπιστώνουμε ότι μέδουσες αυτές ε, παίρνουν τα ΟΑ Ξεκινήσαμε μία έρευνα, ελπίζουμε να έχουμε χρηματοδότηση, γιατί θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε ένα μάστερ που κάνουμε τις επιπτώσεις της μέδουσα στον πληθυσμό του ερυθρού τόνου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έχουμε από το 2009. Κάθετα βλέπετε τον όγκο των ΟΟΝ σε καθημερινή βάση. Δεν φαίνονται καλά κάτω τα νούμερα, αλλά είναι οι ημερομηνίε από 23 Μαΐου του 2009 μέχρι τις 20 Ιουλίου του 2009. Διαπιστώνουμε ότι γύρω στις 9 Ιουνίου ξεκινάει το μοντέλο αναπαραγωγής. Φαίνεται ακόμα και η ώρα ανάμεσα στις 2 και στις 3 ή 3 με 4 καμιά φορά και 4 με 5 το 2010 είχαμε το ίδιο μοντέλο λίγο πολύ επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα σας τα πω σύντομα ξεκίνησε η αναπαραγωγή για την ομάδα αυτή ομάδα ε, ήταν ομάδα η οποία πρώτη φτάνει στο χώρο ε, αλίευσης Όταν ξεκίνησε η αναπαραγωγή αυτού της ομάδας ήρθανε κι άλλοι, ε? Είναι η πρώτη πρώτη, Τόνι. Το 2010 ξεκίνησε μια εβδομάδα νωρίτερα η αναπαραγωγή, παρόλο που η θερμοκρασία ήταν ίδια. Εδώ προσπαθώ να σας εξηγήσω, το βλέπετε, σε καθημερινή βάση τι έγινε και προσπαθούμε να δούμε εδώ ποιο είναι το ποσοστό που φτάνει κάθε μέρα. Την πρώτη μέρα, 9 Ιουνίου, έχουμε το ποσοστό που φτάνει που είναι 1%. Γύρω στις 13 Ιουλίου πάντως και τις δύο χρονιές φτάνουμε στο 100% για την ομάδα αυτή. 13 Ιουλίου δηλαδή είναι και για τις δύο ομάδες. Τι συμπέρασμα βγάζουμε. Ότι η περίοδος που δεν γίνεται λήψη είναι 15 Ιουλίου. Μερικές φορές ε, είναι και λίγο νωρίτερα όπως έγινε το 2010. Ήταν 8 Ιουνίου βλέπουμε ότι η αλία γίνεται πριν λάβει χώρα αναπαραγωγή του τόνου. Δηλαδή εμείς παίρνουμε δείγματα από τη θάλασσα που έχουν αναπαραχθεί και είναι το 10 με 15% της δυνατότητας που υπάρχει. Κάναμε και έναν υπολογισμό Ποιος είναι ο αριθμός? Το 2010 βάσει της ισπανικής ποσόστασης. Της ποσόστασης που είχε η Μπαλφεγό, που είχε η Φουέντες, βάσει όλων αυτών αποφασίστηκε το βάρος και καταλήξαμε σε μισό εκατομμύριο γόνους. Σας εξηγώ με ποιο τρόπο γίνεται η αναπαραγωγή. Ποιο είναι το μοντέλο της παρουσίας αναπαραγωγής, ειδών αναπαραγωγής. Εξαρτάται πάντα βέβαια από το ποσοστό αλίευσης, βδομάδα, τη βδομάδα, από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο για να δούμε πότε έχουμε την μέγιστη απόδοση. Δηλαδή πότε υπάρχει πιο έντονη δραστηριότητα. Και είναι αυτή. Και πάλι εσείς δεν βλέπετε τις ημερομηνίες, είναι 18 με 19 Ιουνίου. Τι έχουμε εδώ. «18 με 28 Ιουνίου» το χρόνο πώς είναι το μοντέλο αυτό. Επίσης είναι γύρω στις 18 με 30 Ιουνίου. Τι επιπτώσεις έχει αυτό. Όταν λέμε ότι 15 Ιουνίου εμείς λέμε ότι σταματάει η αλίευση. Και μιλάμε πάντα για τις βαλαρίδες νήσους αποκλειστικά και μόνο, έτσι. Έχουμε τα δείγματα αλλά μόνο τα δείγματα. Αφήνουμε να γίνει παραγωγή χωρίς κανένα εμπόδιο. Μερικές φορές δεν υπάρχει πλούτος αλλιεύματος. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν φυσικά την παρουσία. Είμαστε στην Μεσόγειο, έτσι η περίοδο απαγόρευση αλίευση είναι ίδια για όλη την Μεσόγειο. Όμω, ένα μήνα νωρίτερα αρχίζουν τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο από ό,τι στη Δυτική. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά φάσματο. Το λογικό θα ήταν ότι οι περίοδοι απαγόρευση αλίευση να προσαρμόζονται στη συμπεριφορά των, ε, της αναπαραγωγής. Να υπάρχει προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Την ενημέρωση την έχουμε, την πληροφορία την έχουμε. Θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και στην πράξη. Εδώ βλέπετε ετησίως τα αλλιεύματα και τα ποσοστά ε, κιλά ανά ημέρα. Βλέπετε τη λευκή γραμμή που δείχνει ότι 2009 και 2010 βλέπουμε μια έντονη δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να δείχνει, αν το προσέξετε καλά, μέχρι τις ημερομηνίες 8 Ιουνίου, 9 Ιουνίου, πότε τελικά ολοκληρώθηκε η αλίευση. Η μείωση δείχνει την αλίευση όταν υπάρχει χαμηλότερη δραστηριότητα. Ο δείκτης αυτός κιλά την ημέρα δείχνει ποια είναι η κατάσταση στις 8 Ιουνίου. Αλλιώ υπάρχει κίτρινη γραμμή. Είναι θετικές τάσεις οι οποίες θα έπρεπε να βοηθήσουν να υπάρχει μικρότερη αβεβαιότητα. Γιατί έτσι βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις που επικρατούν. Στο Μαρόκο, στην ε, Ισπανία, ε, στη Γαλλία και έχουμε και στοιχεία και για την Ιαπωνία ακόμα. Όλοι, όλες αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στα επιστημονικά ε, στοιχεία, αυτά που σας δίνω. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Γορδό, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Σίγουρα θα υπάρχουν μετά ερωτήσεις. Συνεχίζουμε. Πάντα από την επιστημονική κοινότητα το λόγο έχει ο κύριος Δεγκουάρα, που είναι επιστημονικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. ¿Quieres, quieres, quieres,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 Uh, Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στην στο επιστημονικό υπόβαθρο σε σχέση με την αποθέματα ε, ε, μετά από θέματα του ερυθρού τόνου, του Ατλαντικού, με βάση και τις εκτιμήσεις Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΚΑΤ. Following the, uh, λοιπόν αποθεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή της ICAT. Σημειώνονται σημαντικές θετικές εξελίξεις ως προς τα αποθέματα του ερυθρού τόνου Ανατολικού Ατλαντικού σε σύγκριση με την αρνητική κατάσταση που είχε καταγραφεί από την προηγούμενη μελέτη το 2008. Εν ώψη της συνεδρίασης ΙΤΕΣ της ΔΟΧΑ, της Διεθνούς δηλαδή Σύμβασης για την Προστασία των Απολυμμένων Ειδών. Και βάσει της οποίας το 2010 κατέθεσε οι ΣΥΤΕΣ τις εκτιμήσεις της. Προηγούμενες λοιπόν εκθέσεις, τις SCRS, ζητούσαν ε, την εισαγωγή νέων μέτρων, έκροναν τον κόδωνα του κινδύνου, ασκούσαν σαφείς πιέσεις μεταξύ άλλων για περιορισμό της ελευτικής δυνατότητας, χρονικό περιορισμό των, ε, του, της αλλιεύσης, μέχρι και πλήρη απαγόρευση ε, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, σημαντική μείωση των επιπέδων των ΤΑΚ. Βλέπουμε λοιπόν από τη συνολική, το συνολικό μήνυμα που, που αποστέλει η αξιολόγηση αποθεμάτων του 2010 ότι βελτιώνεται η κατάσταση και με 13.500 ε, τάκ εκατομμύρια τόνους ε, εξακολουθεί να βελτιώνεται το απόθεμα ερυθροτόνου. Πλην όμως και παρά τα θετικά σημάδια αποφασίζει στις 2010 η ΚΑΤ την εισαγωγή νέων μέτρων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται το 2011, πέρα δηλαδή της επιπλέον μείωση των ε, ΤΑΚ και επιπλέον η Επιτροπή Συμμόρφωσης λαμβάνει περισσότερες εξουσίες για να προσδιορίσει το κατά πόσον μπορεί μία CPC να ε, ορίσει ή όχι αλληλευτικές δυνατότητες. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στα δεδομένα πριν από τις συνεδρίες του, της ΣΥΤΕΣ του 2010 για να σημειώσουμε ότι καταρχάς τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η SCRS, η Επιστημονική Επιτροπή, η ΚΑΤ, ε, περιορίζονταν στα δεδομένα μέχρι το 2006 μόνο. Δεδομένα που πήγαν στην ΣΥΤΕΣ το 2010. Διότι ναι, έγινε η μελέτη 2008, αλλά δεν υπήρχαν δεδομένα για το 2007 καθόλου. Και άρα τα στοιχεία που συμπεριέλαβε στη μελέτη τη ΕΣΥΑΡΕΣ αφορούσαν μόνο την περίοδο μέχρι 2006. Και όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, υπολογίστηκε συνολικά σε 80.000 μετρικούς τόνους το συνολικό απόθεμα του ερυθρού τόνου Ανατολικού Ατλαντικού. Ωστόσο, όπως είπαμε, άλλαξε δραστικά η κατάσταση και κυρίως διότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση έφταναν μέχρι και το 2009. Έτσι, με τις επιπλέον πληροφορίες που δόθηκαν, με τα νέα στοιχεία, με τις ε, ε, αλλαγές και τα μέτρα όπως περιορισμό των ΤΑ και της περίοδου αλίευσης ή την αύξηση των ε, ε οφθαλμών δείχνουν μια σημαντική αύξηση με βάση την ανάλυση του 2010 κατά περίπου 180.000 μετρικούς τόνους, δηλαδή 75% των υψηλότερων ε, αποθεμάτων ερυθρού τόνου που έχουμε σημειώσει στην ιστορία. Οι δείκτες λοιπόν που οδηγούν προς τη βελτίωση αυτή είναι δείκτες και από τα αλλιεύματα ε, ε, των Ισπανικών υδάτων και των Μαροκινών και στο κάτω μέρος της Καμπύλης βλέπετε ότι υπάρχει, έτσι βελτίωση. Για τα ε, ιαπωνικά σκάφη επίσης στον Ανατολικό Ατλαντικό σημειώνονται θετικές εξελίξεις, έχουμε θετική τάση. Ενδείξεις που έχουν να κάνουν με τα αλλιευόμενα ψάρια επίσης σημειώνουν σημαντική αύξηση περί το 2008-2009 και διότι ε, αυξήθηκε το ελάχιστο μέγεθος, δηλαδή ο κανόνας του ελάχιστου μεγέθους, αλλά και λόγω άλλων μέτρων που εισήχθηκαν. Έτσι, μελέτες τοπικού χαρακτήρα ε, που είχαν πραγματοποιήσει οι γαλλικές κυρίως ε, υπηρεσίες στην περιοχή και βλέπετε τις γεωγραφικές περιοχές την περίοδο 2002-2003 δείχνουν μια διαφορά στον αριθμό των κοπαδιών τόνου που σημειώνονται σε αυτή την περιφερειακή ε, μελέτη και σε σύγκριση με τα τωρινά στοιχεία διπλασιασμό των κοπαδιών, κυρίως δεν των νεαρών ηχθείων. Σημαντική αύξηση του πληθυσμού νεαρών ηχθείων. Η GPYP, το πρόγραμμα δηλαδή ε, έρευνας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΑΤ, είχε υπολογίσει ελάχιστο ε, κατεκτήμηση βάρος ε, στους 18.000 μετρικούς τόνους κατά προσέγγιση αλλά αν κοιτάξουμε τις περιοχές όπου έγινε η έρευνα, οι 4 και οι 5, οι 4 δηλαδή η Λιβύη και οι 5 η Αίγυπτος, πραγματικά δεν είχαν ερευνηθεί και άρα δεν περιεχόνταν τα στοιχεία τα σχετικά. Η Κροατία επίσης στην, επίσημη, στην επίσημη έκθεση της προς την ΕΚΑΤ για τον ε, ερυθρό τόνο και τα μικρά πελαγικά είδη για το 2010 για την αληφτική περίοδο σημειώνει υψηλότερη συγκέντρωση νεαρών ηχθείων και, και ενηλίκων ε, ηχθείων στην περιοχή της Ανδριατικής. Και σημειώνονται και ε, παρουσία ψαριών σε περιοχές που δεν είχε προηγουμένως εμφανιστεί ε, το ψάρι αυτό ή σε πολύ ψηλότερα σε πολύ ψηλότερη συχνότητα. Φερρυπίν, Μάλτα. 2009-2010 ερυθρός τόνος σε χιλιάδες ε, ατόμ, άτομα, σε ομάδες χιλιάδες ατόμων απελευθερώθηκε από κλοβού στο Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία. Και έτσι η Επιστημονική Επιτροπή της ΙΚΑΤ υπολογίζει ότι τα αλλιεύματα ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τα, βελ, με τα υψηλότερα αποθέματα, τα υπολογιζόμενα υψηλότερα αποθέματα, ήταν στην πραγματικότητα χαμηλότερα από τα καταγραφέντα. Και έτσι δηλώνει ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αγνωρίζει όμω ταυτόχρονα η Επιστημονική Επιτροπή ότι πιστεύει πω οι στόχοι τη ΙΚΑΤ μπορούν κατά τρόπο αιφόρο να εξασφαλιστούν με το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης και ακόμη και με επίπεδο ΤΑΚ στο ύψος των 13.500 εκατομμυρίων τόνων. Και μπορούσε ε, να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη απόδοση σε ύψους 50.000 περίπου μετρικών τόνων. Επίσης εξετάστηκε κατά πόσον οι στόχοι της ΣΥΚΑΤ έχουν ε, επιτευχθεί ή όχι, ανάλογα με τους στόχους που είχαν προσδιοριστεί σε περίπτωση, στην περίπτωση του κάθε έτους. <coughs> Θα δείτε στο γράφημα ότι έχω σημειώσει το 13.500 ε, μετρικούς τόνους με πιθανότητα για το 2022 κατά 63% να επιτευχθεί αυτός ως στόχος. Επίση, σε προηγούμενε εκθέσει η Επιστημονική Επιτροπή είχε δώσει μεγάλη συμφωνία, σημασία σε στρατηγικέ ε, διαχείριση ε, με την χρήση του αποκλεισμού μερικού ή κατά την περίοδο της οτοκίας ε, για το 2010 και βλέπουμε ότι μερικός αποκλεισμός ήδη έχει ξεκινήσει ενώ έχουμε μόνο ε, ενός μηνός διάρκεια δυνατότητας αλίευσης με το γρηγρή, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με πλήρη αποκλεισμό ε, της ε, περίοδου, με πλήρη απαγόρευση δηλαδή για την περίοδο της ε, οτοκίας. Στη συνέχεια βλέπετε στον πίνακα τους, ε, ε, την κατανομή για τον ερυθρό τόνο της, ε, τα πάλι στο 13.500 μετρικούς τόνους με ποσοστό, με πιθανολόγηση ότι θα επιτευχθεί ο στόχος κατά 0,91% ε, ήδη το 2015, άρα πιο θετικές ακόμη οι προβλέψεις. Επίσης έχει προβλέψει και άλλα μέτρα η ΚΑΤ. Έχουμε παρατηρητές πάνω στα σκάφη, έχουμε άσκηση πιέσεων ε, για την αξιολόγηση του ε, βάρους των παράπλευρων αλλιευμάτων, των παρεμπιπτόντων αλλιευμάτων κ.ο.κ. Έχουμε πίεση για την παρουσίαση ενός σχεδίου αλλίευσης και προς την Επιτροπή Συμμόρφωσης. Μια μελέτη, που, μια συνεδρία μάλλον πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελόνη του προηγούμενο μήνα και όπου τα κράτη παρουσίασαν τα αλληλευτικά τους προγράμματα, σχέδια, τα οποία θα εγκριθούν μόνο εφόσον επικυρωθούν από τις αντίστοιχες ε, CPCs ε, και από τις άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι για τον αριθρό τόνο στον, ε, Ανατολικό Ατλαντικό 12.900 επίσημα τα στοιχεία για τον ερυθρό τόνο Στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 12.899 12 μετρικούς τόνους, ε, από τους οποίους όμως θα πρέπει να βγάλουμε για τους γνωστούς λόγους στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Άρα πέφτουμε περίπου ε, στους 12.000, στους 12.000 περίπου μετρικούς τόνους με την ε, διαγραφή από τον κατάλογο των κρατών που παρουσιάζουν αυτές τις σχολές στην εποχή. Επίσης, σημειώνεται ότι ήδη έχουν τα ηχθειοτροφία συμβάλει σημαντικά με τα, ε, με πειράματά τους ε, για αναπαραγωγή, με το γενετικό υλικό, με, τις, ε, με τη συμμετοχή σε διάφορα πειράματα σημαντικά στην διατήρηση και ενίσχυση των αποθεμάτων. Γίνεται συζήτηση για ανάπτυξη, για την ορίμανση του ζώου μέσα στα, στο ηχθειοτροφείο, σε κλοβούς, βελτίωση των συνθήκων κράτη σε κλοβούς και για να ολοκληρώσουμε ε, ο κλάδος της εκτροφής δείχνει βούληση να στηρίξει τις επιλογές της ΑΕΚΑΤ με βάση επιστημονικά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε ε, διατήρηση και βελτίωση των αποθεμάτων του ερυθρού τόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δεγκουάρα, αυτά τα τελευταία που μας είπατε δείχνουν ότι υπάρχουν ελπίδες για ανάκαμψη. Υπάρχουν τέτοια δείγματα ήδη. Επιβεβαιώνεται αυτό από αυτά που μας είπατε κι εσείς. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Μιέλγκο έχει το λόγο, ο οποίος θα μας μιλήσει εκ μέρους μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων. Ποια είναι η θέση της ε, World Wide Fund και της Greenpeace. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Έχω αλλάξει κάπως τη σημερινή μου παρουσίαση την τελευταία στιγμή. Δεν γινόταν και διαφορετικά, γιατί τα τελευταία γεγονότα στη Λιβύη, που είναι κύριος χώρος αλίευσης ε, ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο, όπως επίσης και η φυσική αλλά και πυρηνική καταστροφή στην ε, Ιαπωνία, όπου επίσης έχουμε πολύ μεγάλη αλίευση ερυθρού τόνου και παράλληλα η απαγόρευση που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ερυθρό τόνο τροποποιούν καθοριστικά θα έλεγα η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την δραστηριότητα εκτροφής και αλίευσης του ερυθρού τόνου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σήμερα, κατά την γνώμη μου, η συνάντηση αυτή έχει να κάνει με έναν τομέα και ένα κλάδο που κατά τη γνώμη μου ε, ξεκίνησε με σοβαρά προβλήματα ήδη από το 2008 Εννοείται ότι διαφωνώ με πολλά από όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Θα τα δούμε όμως σε λεπτομέρειες. Θα επικεντρωθώ πιο συγκεκριμένα στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, 2008, 2009 και 2010, τόσο όσον αφορά την ε, ανιχνεσιμότητα, δηλαδή το περίφημο Bluefin Tuna Catch Document που είναι ένα σύστημα ε, ανιχνευσιμότητας, ιχνηλασιμότητας ε, του ερυθρού τόνου. Είναι ένα σύστημα που λέει ότι για κάθε αλίευση υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο συνοδεύει το είδος από τη στιγμή που αλλιεύεται μέχρι τη στιγμή που φτάνει στον τελικό του προορισμό. Κυρίως στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία το έφτιαξε αυτό, αλλά ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Κορέα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε λοιπόν τα τρία τελευταία χρόνια με αυτό. Τα νούμερα που μας φτάνουν δεν ε, είναι θετικά. 2008, 2009 και 2010 διαπιστώνουμε από τις βάσεις δεδομένων που έρχονται από τα Ιαπωνικά ή Αμερικανικά τελωνία, αλλά και τα στοιχεία που μας έρχονται από βάσεις δεδομένων ε, της Eurostat, για να έχουμε μια ιδέα το ποιες είναι οι ροές, οι εμπορικές ροές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρέει ο πίνακας που δείχνει σε μπλε τις, κολ, τις στήλες που έχουν να κάνουν με την εμπορία του τόνου που, που αλλιεύτηκε τη συγκεκριμένη χρονιά, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, γιατί πουλιέται κατευθείαν στην Ιαπωνία, οπότε δεν εξάγεται. Ούτε συμπεριλαμβάνονται χώρες όπως είναι η Κίνα, η Κορέα και τα Ιωάννη. Στην πράξη δηλαδή, αυτός ο ερυθρός τόνος είναι από τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και την Μεσόγειο και έχει να κάνει μόνο με τις χώρες που βρίσκονται στην περιοχή. Στην κόκκινη στήλη βλέπετε τις δηλώσεις αλίευσης από τις ίδιες αυτές χώρες. Πώς δήλωσαν στην ΙΚΑΤ. Από το 2008 δηλαδή τα συμβαλόμενα μέρη στην ΙΚΑΤ δηλώνουν εβδομαδιαία και μηνιαία τα ελιεύματά τους. Εμείς πήραμε τα μηνιαία στοιχεία γιατί θεωρούμε ότι είναι τα πιο πλήρη. Και έτσι καταλήξαμε στην ετήσια αλίευση και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορές ανάμεσα στην πραγματικότητα που έχουμε από το εμπόριο και την πραγματικότητα που έχουμε από τι δηλώσει αυτές αλλίευση. Όταν όμως πάμε στη βάση των στοιχείων του συστήματος, βλέπουμε στις πράσινες στήλε τα κιλά, σε κιλά, έτσι, τις ποσότητες που έχουν αλλιευθεί και έχουν περάσει μέσα από το σύστημα ανείχνευσης του ερυθρού Από το 2008 φαίνεται έτσι ότι υπάρχει μείωση των αλλιευμάτων γιατί υπάρχει χαμηλότερη αλίευση, λιγότερη αλίευση και πιο περιορισμένος χρόνος ε, κατά τη διάρκεια του οποίου επιτρέπεται η αλίευση. Απ' την άλλη υπάρχει αύξηση στη διαφορά ανάμεσα στο δηλωθέν αλίευμα βάσει των αιτήσεων δηλώσεων η βάση του εγγράφου αυτού του BCD και των ποσοτήτων που όντως φτάνουν στο εμπόριο. Οι μπλε στήλε δεν περιλαμβάνουν, όπως ε, σας έχω πει, τον μεταπημένο τόνο. Αλλά αναφέρουν τον άγριο τόνο. Πώς γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν ε, πολλοί και διάφοροι παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε ποια είναι τα ποσοστά πάχυνσης. Έχουμε την επίσημη πάχυνση που έχουμε από την ΙΚΑΤ και που εγκρίνει η ΙΚΑΤ το 2009 στο Ρεσίφε ήταν που αποφασίστηκε, στοιχεία τα οποία βέβαια είναι σε αντίθεση με κάθε επιστημονική λογική. Γιατί δεν είναι δυνατόν σε εξημένες να έχουμε πάει σε 200%. Κανένας δεν θα το πιστέψει αυτό. Ο πίνακας αυτός που έχετε εδώ στα αριστερά έτσι λέει. Και από την άλλη Έχουμε παράδειγμα μια επιχείρηση για την οποία έχω δουλέψει, από που φαίνεται ανακλωβό πάχυνση και αναβάρος ε, ψαριού στο τέλος της περίοδου αλίευσης. Αλλά και εδώ πάλι αν υπάρχει κάτι λογικό είναι καθαρά θέμα σύμπτωσης. Γιατί δεν υπάρχει λογική εδώ. Οπότε θα έπρεπε να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα αυτό της πάχυνσης. Πρόκειται για science fiction. Έχουμε όμως και κάτι άλλο. Ότι δεν δηλώνονται αλλιεύματα. Εδώ έχετε έναν, ε, μια ανακεφαλαίωση στον πίνακα αυτό και πρόκειται για τον τόνο ο οποίος έχει μεταφερθεί ο οποίος έχει εντοπιστεί τη στιγμή της εκφόρτωσης βάσει στοιχείων του ΙΚΑΤ, e του εγγράφου αυτού ανείχνευσης. Μετράμε δηλαδή την ε, δήλωση, ας πούμε ότι έχουμε 100 τόνους από χίλιους αλείς στον τάδε κλοβό στο τάδε μέρος της τάδε χώρας και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν κάποιος δει τα στοιχεία της εκφόρτωσης διαπιστώνει ότι αυτοί οι χίλιοι έγιναν 2.000 οι οποίοι αλλιεύσαν 300 ε, τόνους. Όσο και αν θέλετε να με πείσετε, ε, αφού έχει αλλιευθεί το ψάρι δεν μπορεί να μεγαλώσει πια. Και πάω και ακόμα πιο μακριά προσέτουμε και, έναν, και μια άλλη κολόνα για το ίδιο μέρος. Αναφέρεται ότι υπάρχει το ψάρι που πιάστηκε μια συγκεκριμένη χρονιά, την επόμενη χρονιά είναι 100 ε, τόνοι παραπάνω. Μα πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Το 2008 έχουμε τον αριθμό περιπτώσεων που δεν έχουν δηλωθεί ως μεταφορά ζώντος ηθιος. υπάρχουν 8 περιπτώσεις το 2009 και 0 το 2010. Δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση γιατί, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η περίοδος. Ούτε αλίας, ούτε της ε, δήλωσης που γίνεται το 2011 και το 2010. Και η περίπτωση των περιπτώσεων που δεν δήλωσαν την μεταφορά το 2008 1η Μαρτίου έχουμε 26 περιπτώσεις που σημαίνει ότι δεν έχουμε στοιχεία για το 2008 σε 26 περιπτώσεις. 25 το 2009 και 18 το 2010. Αλλά και εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι ίσως θα έπρεπε και εδώ να μπει 0 γιατί είναι νωρίς, γιατί ακόμα δεν έχουμε όλες τις ε, δηλώσεις για το 2010, δεν έχουν γίνει όλες. Αυτά ισχύουν για όλα τα συμβαλώμενα μέρη όσον αφορά τις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο. Αλλά έχουμε τρεις περιπτώσεις μεταξύ πολλών άλλων, από τρεις χώρες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο παράδειγμα. Κράτος μέλος, θα το ονομάσουμε Α. Εκεί για το 2008 έχουμε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία που ανακοινώνονται βάσει του BCD για ατομικά και για τόνους που μεταφέρονται. Διαφορά λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία έχουμε πάρει από το ίδιο το Υπουργείο Αλίας της εν λόγω χώρας Α. Ελέγξαμε δηλαδή τα στοιχεία BCD και τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο της συγκεκριμένη χώρας Α και διαπιστώνουμε ότι το 2008, σύμφωνα με το Υπουργείο, είχαμε 36.726 περιπτώσεις, ενώ βάσει των στοιχείων της ΙΚΑΤ έχουμε 32.770 περιπτώσεις. Έχουμε Επίσης, δηλωμένες περιπτώσεις στο ΙΚΑΤ 151, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο ήταν 177. Και βλέπετε και τη διαφορά μετά. Άρα δεν γνωρίζουμε τι έγινε με 342, με 342 τόνους. Δεύτερο παράδειγμα, άλλη χώρα μέλος, Β ας την ονομάσουμε. Εκεί έχουμε μεγάλες διαφορές ανάμεσα για το 2009 των αλλιευμάτων των δηλωμένων βάσει στοιχείων BCD και τα δεδομένα από το logbook της ε, αρμόδιας για την αλληλεία αρχή της συγκεκριμένης χώρας Β. Από το logbook της χώρας ε, αυτής έχουμε αρκετά πλήρη στοιχεία πολλά στοιχεία. Δεν χρειάζεται να σας τα αναφέρω εδώ. Το κράτος μέλος λοιπόν, αυτό το 2009, είχε 3.196, ενώ βάσει των δεδομένων της ίδιας της δικιάς του ελευτικής χαρτής είχε 3.509 τόνους. Δήλωσε όμως αλίευσε 3.509 τόνους όταν κάνουμε ε, τη διασταύρωση. Βλέπουμε 2.451 τόνους βάσει του logbook. Του logbook. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί αλλιεύματα στα logbooks των ε, σκαφών που δεν αναφέρονται στη βάση δεδομένων BCD. Τρίτη περίπτωση. Και με αυτήν θα τελειώσω. Παράδειγμα μιας χώρας μέλος, γάμα, ας την πούμε, όπου υπάρχει δραστηριότητα πάχυνσης παράνομη. Και γιατί παράνομη. Γιατί δεν έχει καταγραφεί στην ΙΚΑΤ η δραστηριότητα αυτή με άδεια για πάχυνση. Που σημαίνει ότι πρόκειται για θέμα του ανταγωνισμού. Μας εξήγησαν στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης της ΣΥΚΑΤ ότι ε, μπήκε και ο τόνος με τα ποσοστά πάχυνσης εντοπίσαμε 167 είδη που 26-27 τόνοι βρίσκονται στην εμπορία στην Ιαπωνία μπήκαν 610 τόνοι ζωντανού τόνου. Βέβαια, εύκολο είναι άμα δεν ξέρει κανείς τι λένε, ότι το πρώτο βράδυ έφυγε, ξέφυγε. Για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, είναι 12 εκατοστά το μάτι του δικτυού. Και έτσι θεωρητικά έφυγε, ξέφυγε, τόσκασε ο τόνος. Μα είναι δυνατόν να βάλεις ε, τέτοιες ποσότητες μέσα σε ένα κλωβό. Εδώ μιλήσαμε πολύ και θα τελειώσω με αυτό κυρία Πρόεδρε. Μιλήσαμε πολύ για τα αποθέματα. Πρέπει να ξέρετε το εξής. Ότι το Συμβούλιο CSFR συζητάει πολύ για το μέγεθος και παίρνει αποφάσεις ιστορικής σημασίας. Πρώτον, τι γίνεται στην Ιαπωνία. 20 χρόνια, 122.000 περιπτώσεις έχουμε. Στην Ισπανία επίσης. Και τέλος στη χώρα των Βάσκων. Τρεις διαφορετικές κατηγορίες σκαφών. Σήμερα, να ξέρετε, ότι δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε για τα λιεύματα μέσα στην ε, Μεσόγειο. Και συνεπώς, η γνώμη μου είναι ότι, και συμφωνούν σε αυτό και πολλοί άλλοι, ότι εδώ η επιστημονική προσπάθεια που γίνεται θυμίζει βουντού. Γιατί δεν ξέρουμε για τα γρηγρή, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Ναι, λένε πολλοί, υπάρχει μια βελτίωση όσον αφορά τις βαλαρίδες μόνο. Και θα συνεχίσω, διακόπτη πρόεδρος, ολοκληρώστε και τελείως δεν θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Έχουμε μισή ώρα, το έτσι καλώς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Συνεχίζω μιλητής. Έχουμε αναλύσει τα στοιχεία της αγοράς για όλων των ερυθροτόνο της Μεσογείου που πουλιέται από το 2002 μέχρι, από το 2001 μέχρι το 2009 στην ικτιός, στις Ιαπωνία. της Ιαπωνίας. Τα στοιχεία για την επόμενη χρονιά θα τα έχουμε σε λίγους μήνες στη διάθεσή μας. Τα ποσοστά λοιπόν αντιστοιχούν στα 120 κιλά και παραπάνω που πουλούνται στις ηθιόσκαλες αυτές όλα αυτά τα χρόνια. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αύξηση των ποσοστών. Το 2008 μάλιστα ήταν τραγική χρονιά και βλέπουμε ότι υπάρχει μια κάποια βελτίωση το 2009. Αν έπρεπε να αναλύσουμε τα στοιχεία του 2009, η πλειοψηφία κατά το 95% όχι και παραπάνω είναι από τις Βαλεαρίδες. Στην υπόλοιπη Μεσόγειο τραγική κατάσταση. Και όλα τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε για το 2010 και που φτάνουν στην Ιαπωνία, σε πληστερισμό εκεί, δείχνουν ότι η τάση αυτή συνεχίζεται και συνεχίζεται ιδιαίτερα για τις Βαλεαρίδες νήσους. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιέλγο. Όλες οι παρεμβάσει ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Τώρα δεν ξέρω ποιο θέλει το λόγο. Τώρα έχουμε συζήτηση. Ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους βιρογνώμονες που ήρθαν εδώ σήμερα για τις απόψεις που μας μετέφεραν. Και μια που είναι εδώ, θέλω να τους κάνω κάποιες ερωτήσεις με την άδειά σας. Στον κύριο Απόστολο, δεν θυμάμαι το επιθετό του, λέει ο θέλω να ρωτήσω τα εξής. Για τις επιπτώσεις που έχουν αυτά που συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Ανησυχούν τα πράγματα ένα τμήμα του κλάδου. Ότι τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ιαπωνία επηρεάζουν την κατάσταση, την αγορά και τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Το λαμβάνουν υπόψη τους μελέτες. Έπειτα, Ακούστηκε κάτι ενδιαφέρον για τα αποθέματα και για την αποκατάσταση. Το 80% πιστεύει ότι είναι αρκετό. Ενώ οι εγγύσεις για την αποκατάσταση των ειδών είναι πολύ χαμηλές. Τώρα για τους φίλους, γιατί τους λέω φίλους γιατί πολλές φορές έχουμε βρεθεί και θα ξαναβρεθούμε από την Παλθέγο. Θέλω να ρωτήσω για την καινοτομία, για τον καινοτόμο χαρακτήρα τους να μας μιλήσουν. Να πάνε λίγο πιο πέρα από την καθαρά εμπορική τους δραστηριότητα. Και εντάξει για την Παλθέγο, αλλά για τον τομέα, τον ευρύτερο έτσι όπως οργανώνεται η δραστηριότητα. Η ερώτησή μου είναι και για την Παλθεγό, αλλά και για τον κύριο Μιέλγο. Συμφωνούμε ότι το πρόβλημα σήμερα είναι λίγο είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή αξιοπιστία στα συστήματα ελέγχου στο σύνολο της αγοράς. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη ελέγχου των στοιχείων. Συμφωνούμε ότι υπάρχει γενικά το πρόβλημα, είτε κάνουν καλά τη δουλειά τους είτε όχι. Το θέμα είναι με τους μηχανισμούς και τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά. Και να εκφράσω και μια ανησυχία για την κυρία Γκορδόα, για τις μέδουσες. Και συγγνώμη αν πω κάτι λάθος. Απ' την άλλη μεριά αποτελούν και τροφή για τον τόνο. Έτσι δεν είναι. Οπότε δεν ξέρω τελικά μια τέτοια κατάσταση είναι πιο επώδυνη. Γιατί τόνοι τρώνε τις μέδουσες, αλλά οι μέδουσες τρώνε τα αυγά των τόνων. Μπορεί να μας το αναλύσει αυτό περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Αντρές Βαλέ το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες για αυτά που μας είπαν. Συγχαρητήρια στην Παλθεγό. Από ό,τι φαίνεται η καινοτομία και η τεχνολογία Είναι πράγματα που χρησιμοποιούν για την ε, αποκατάσταση του τόνου. Πολύ καλό. Ο τελευταίος ομιλητής μας είπε ότι δεν υπάρχει αποκατάσταση. Θα μπορούσε να μας πει περισσότερα για την αποκατάσταση, πώς ακριβώς έχει. Έπειτα ο δεύτερος ομιλητής καταδίκασε επανελειμμένα την παράνομη ελεία εκεί είπε ότι πρέπει να καταγγέλλεται. Τι δραστηριότητες έχουν αυτοί για να καταγγέλουν Και τι γίνεται όταν καταγγέλλονται τέτοιες περιπτώσεις. Στην κυρία Άννα Γκορδό. Αυτά που είπατε τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα που είπατε ότι από 15 Ιουνίου σταματάει ματάει περίοδος αλίευσης, αλλά μερικέ φορέ θα έπρεπε να τα νωρίτερα. Ίσως γι' αυτό τα αποθέματα να είναι τόσο χαμηλά, οπότε δεν θα ήταν μια καλή πρόταση να μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις στις δύο αυτές πλευρές της Μεσογείου, η κυρία Λουβίν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρα και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι παρουσιάσεις. Μία ερώτηση προς τον κύριο Σιμεών Ντεγκουάρα. Αν κατάλαβα καλά, εκπροσωπείτε την Ένωση Διεκτοκαλλιέργειας. Θα ήθελα να ακούσω λίγο παραπάνω για το ποιους εκπροσωπείτε γιατί μου έκανε εντύπωση, είσαστε πάρα πολύ σαφής και πιστικός όσον αφορά ε, την ε, εξέλιξη των αποθεμάτων τα τελευταία χρόνια. Στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε την κατάσταση των αποθεμάτων για τον ερυθρό τόνο πριν από έξι μήνες. Και τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάσατε είναι ιδιαίτερα πιστικά. Ε, λέτε ότι υπάρχει μια ανάκαμψη των αποθεμάτων αν κατάλαβα καλά, οι επιστήμονες ε, έχουν, ε, πιστεύουν σε διαφορετικά σενάρια όσον αφορά τον υπολογισμό των αποθεμάτων. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ε, με τους επιστήμονες. Εγώ είμαι βέβαια πιο εξοικειωμένη με τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά οι επιστήμονες μας δίνουν διαφορετικά στοιχεία. και διαφορετικά στοιχεία τοποθετούν στα διάφορα μοντέλα εκτίμησης και αξιολόγησης των αποθεμάτων. Επομένως, ρωτώ πόσο σίγουρα είναι τα στοιχεία που μας δίνετε εσείς ε, για τα διάφορα σενάρια και ποιος εγγυάται τα νούμερα, τα δεδομένα αυτά τα οποία αναφέρατε. Επίσης, αναγνωρίζω το γεγονός ότι η βιομηχανία, ο κλάδος μας λέει ότι όλα τα στοιχεία που μας δίνουν οι επιστήμονες είναι ε, ξεπερασμένα. Αναφερθήκατε στους στόχους το 2006, έχουμε τα στοιχεία μέχρι το 2008, τώρα όμως είμαστε στο 2011. Επομένως, λογικά θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα για μία μείωση των αποθεμάτων ε, από το 2008 και μετά. Ή έχουμε όλες αυτές τις αβεβαιότητες, οι οποίες έχουν ε, ενταχθεί στα όλα στους υπολογισμούς για τον αριθμό των ψαριών που έχουμε. Επομένως, ε, ρωτώ εγώ πόσο αξιολογείται την προσέγγιση ε, την προληπτική. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν κάνουμε τους υπολογισμούς μας ε, και όταν ε, αποφασίζουμε για το τι θα κάνουμε λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε τα στοιχεία μέχρι το 2008 και όχι μέχρι το 2011. Επίση, το μέσο μέγεθο των ψαριών είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση ε, όταν θέλουμε να αποφασίσουμε αν υπάρχει υπεραλία ή όχι. Ο μέσο όρο βάρου και μεγέθου ε, των τόνων ε, δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάκαμψη ή μιλάμε για μικρά μεγέθη, έχουμε νεαρά ζώα τα οποία αλλιεύονται. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Στις 12.30 πρέπει να έχουμε τελειώσει και θέλω να σας δώσω σε όλους το λόγο για να απαντήσετε. Γιατί πράγματι ε, μεταξύ σας είπατε και αντιφατικά πράγματα. Κύριε Κορδό, είπατε ότι υπάρχει πρόοδος στην έρευνα για την αναπαραγωγή σε κλοβούς κλπ. Στην Ανατολική Μεσόγειο η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα πριν από ό,τι στη Δυτική, έτσι δεν είναι. Είναι ένα θέμα γνωστό στην επιστημονική κοινότητα. Πράγματι, δεν είναι λογικό να έχουμε την ίδια περίοδο απαγόρευσης ε, αλίας παντού. Υπάρχει κάποιος άλλος επιστημονικός λόγος ή άλλου είδους που εμποδίζει την ΕΚΑΤ να πάρει μια απόφαση που σε όλους μας φαίνεται προφανής και λογική. Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο με την αντίθετη σειρά για να απαντήσετε και σε αυτά που είπατε μεταξύ σας. Αλλά 12.30 πρέπει να τελειώσουμε γιατί οι πρέπει να φύγουν, λέει ο Πρόεδρος. Συνεπώς είσαστε πέντε, δύο λεπτά ο καθένας. Πρώτος ο κύριος Μιέλγο. Δύο λεπτά, ε, ακριβώς. Και θα χτυπήσω εδώ το σφυρί μου για να σταματήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στον Ευρωβουλευτή Ρομέδα. Η σημερινή καταστροφική κατάσταση στην Ιαπωνία αλλάζει όλα τα δεδομένα. Οι βασικοί εισαγωγείς ενημερώνουν τους κύριους παραγωγούς ερυθρού για το ότι όλα βρίσκονται σε κρεμότητα. Σήμερα το πρωί διάβασα ένα νέο ότι μια σημαντική ομάδα απάχυνσης ε, ισπανική ερυθρού τόνου σταματάει τις εξαγωγές της στην Ιαπωνία. Κάθε γεν που έχει στα χέρια της ιαπωνική οικονομία μην ξεχνάμε ότι θα χρησιμεύσει για την ανοικοδόμηση της χώρας. Και εξάλλου δεν ξέρουμε και πολύ καλά τι θα συμβεί ακόμα στη χώρα αυτή. Και υπάρχει και η Λιβύη όπως σας είπα και όλα δείχνουν ότι ο φίλος πόλεμος στη Λιβύη θα συνεχιστεί. Και δεν θα ήταν σοφό να μεταφέρουμε κλοβούς στην ε, περιοχή αυτή αλίευσης. Παρόλο που σας είπα το 70% ανάλογα βέβαια με τη χρονιά μας έρχεται από εκεί. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Ο κύριος Τεγκουάρα τώρα. πολλές ερωτήσεις για το θέμα της ανάλυσης των δεδομένων και τα διαφορετικά σενάρια, το RCRS και όλα τα, ε, όλοι οι οργανισμοί διαχείρισης της αλίας εξετάζουν τα διάφορα σενάρια με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τελικά ε, επικυρώνουν, αν θέλετε, ή δέχονται τα πιο πιθανά σενάρια είχαν 24 διαφορετικά σενάρια δηλαδή τελευταία φορά που έκανε αυτήν την αξιολόγηση με διαφορετικά στοιχεία που αφορούσαν τα αλλιεύματα και μετά ε, επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα-δύο μοντέλα τελικά τα οποία είναι τα πλέον πιθανά και που οδηγούν στο συμπέρασμα που έχουμε. Έχουμε ε, κάνει την τελευταία εκτίμηση με τα δεδομένα του 2010 και του 2009. Λαμβάνοντα υπόψη και αυτά που έγιναν το 2008 βέβαια. Το 2008 είχαμε στοιχεία που αφορούσαν μονάχα μέχρι το 2006. Τώρα είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε και τα δεδομένα άλλων τριών ετών. Και αυτό άλλαξε αν θέλετε το είδος των δεδομένων που είχαμε. Γιατί η ε, το 2010 η κατάσταση ήταν πλέον πιο σαφής, γιατί είχαμε περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μα. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο γεγονό ότι το 2010 εξετάσαμε ε, το αποτέλεσμα των διαφόρων μέτρων διαχείρισης που είχαν ε, εφαρμοστεί το 2006, 2007, 2008 και το ΤΑΚ περιορίστηκε στα 13.500 τόνους και το ελάχιστο μέγεθος αλίας ε, υπήρχαν στοιχεία, υπήρχαν μέτρα δηλαδή τα οποία ήταν θετικά και οδήγησαν στην ανάκαμψη του αποθέματος. Το 2010 υιοθετήθηκαν περισσότερα μέτρα, εφαρμόσαμε περισσότερους ελέγχους. Είναι επιστημονικά όλα αυτά που σας λέω, αλλά οι δείκτες είναι θετικοί και οι δείκτες υπάρχουν που δείχνουν ότι η τάση θα συνεχιστεί. Έστω και αν η επιστήμονες ε, ανάλογα με το ποιον θα ρωτήσετε μας λένε διαφορετικά πράγματα. Όμως η κατάσταση έχει αλλάξει. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κύριε Γκόρδο. Τρεις ερωτήσεις μου κάνατε. Πρώτα απ' όλα για τις μέδουσες. Και εγώ αναρωτήθηκα το ίδιο πράγμα πριν από μερικά χρόνια. Και ποτέ δεν είχα δει τότε επιστημονικό άθρο. Αλλά μετά είδα ένα τέτοιο επιστημονικό άρθρο. Οπότε έμαθα ότι στη Μεσόγειο μόνο μικρά πελαγιακά είδη έχουμε έτσι στην ε, Μεσόγειο. Ρέγα και λοιπά. Λοιπόν, η διάδοση της μέδουσας στη Μεσόγειο είναι επειδή υπάρχει μείωση του τόνου. Βέβαια δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Από τις πληροφορίες που έχω πάντως αυτό μπορώ να σας πω. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι η μέδουσα που εμείς παρατηρούμε δεν είναι μόνο η ενήλικη αλλά και η μικρή και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην μείωση του τόνου και την μέδουσα. Κάπου επίση, διάβασα πώς στις βαλερίδες ενίσους έχουμε αυτήν την σχέση ακριβώς. Αυτά είναι πράγματα Όσοι δουλεύουν με το πλακτόν το βλέπουν σιγά σιγά και εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους. Είναι ένα θέμα, σας είπα, ήταν η πρώτη ερώτηση που και εμένα μου πέρασε από το μυαλό. Δεύτερη ερώτηση που μου κάνατε. Κατά πόσο τι πρέπει να κάνουμε μάλλον με τα αποθέματα. Πρώτα απ' όλα, Είπατε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Μεσόγειο, όντως όσον αφορά την περίοδο αναπαραγωγής. Εμείς ε, με την έρευνά μας προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι αυτή η διαφορά και αν υπάρχουν γενετικές διαφορές, που δεν υπάρχουν από ό,τι διαπιστώσαμε. Βέβαια με μία ανάμειξη 3% δεν ήταν δυνατόν να απαντήσουμε με βεβαιότητα σε αυτή την ερώτηση περί γενετικών διαφορών. Η τόνοι πάντως που είδαμε στην Ανατολική Μεσόγειο δεν τους βρήκαμε στον Ατλαντικό. Μπορεί να υπάρχει πληθυσμός που είναι κατεστημένος περισσότερο στην Ανατολική ή στην Δυτική Μεσόγειο. Αν οφείλεται στο κλίμα, εντάξει δεν ξέρω, αυτό το λέω έτσι. Και για το τελευταίο. Α, γιατί υπάρχει επιφύλαξη, με ρωτήσατε, επιστημονική για να γίνει διαφοροποίηση στην περίοδο απαγόρευσης ε, αλίευσης στην Ανατολική και τη Δυτική Μεσόγειο. Όχι, άλλος επιστημονικός λόγος δεν υπάρχει, άλλος λόγος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Μπορεί να υπάρχουν ε, προβλήματα σε άλλο επίπεδο, αλλά επιστημονικά άλλος λόγος δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε, ο κύριος Σεράνο. Στην πρώτη ερώτηση του κύριου Ρωμέβα. Χαίρομαι που είπατε ότι είσαστε φίλος μου και εμείς νιώθουμε φίλοι σας. Ε, αναρωτηθήκατε για την αξιοπιστία μας. Εγώ πιστεύω και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή λέει για την ΙΚΑΤ, στην οποία εγώ πιστεύω. Θα φύγετε από την ΙΚΑΤ. Εντάξει αν φύγετε από την ΙΚΑΤ, αλλά όσο βρίσκεστε στην ΙΚΑΤ δεν μπορούμε παρά να έχουμε εμπιστοσύνη στα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε από εκεί. Κύριε Ρωμέβα, τα έχουμε συζητήσει πολύ Δεν είναι δυνατόν να πείτε σε κάποιον ότι οδηγάει καλά, ότι τηρεί τα όρια ταχύτητας, παρόλα αυτά θα του πάρετε το δίπλωμα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται στον τομέα και να μην γίνονται αδικίες. Εμείς ναι, καταγγέλουμε. Καταγγέλουμε συνέχεια και με ονόματα και με επίθετα. Δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι. Εμείς το κάνουμε. Αυτά που ξέρουμε τα καταγγέλουμε στην Επιτροπή Ελέγχου. Και έχουν γίνει πράγματα άλλε φορέ γίνονται πολύ αργά. Εγώ προτείνω να πηγαίνουν επιθεωρητές έτσι στα ξαφνικά. Ο τόνος έχει μια ταυτότητα. Πρέπει οι ελεγκτέ να πηγαίνουν και να τη ζητάνε αυτή την ε, ταυτότητα, να τη βλέπουν. Όσον αφορά για τον κύριο Μέλγο και για τις ε, υπόνοιέ του, για την απαγόρευση εξαγωγών, μα οι αεροπορικές εταιρείες πάνε με ανθρωπιστική βοήθεια και δεν μπορούν να μεταφέρουν τις δικές μας ε, τις εξαγωγές. Φυσικά όμως χρειάζεται τρόφιμα. 16 τόνοι ε, τόνου θα πάνε στην Ιαπωνία σήμερα με ένα αεροπλάνο. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Εξάλλου, κύριε Μιέλγο, λέτε ότι έχετε μελέτη για τους μικρούς ε, τόνους στην ε, ηχθιόσκαλα της Ιαπωνίας. Μα είναι πολύ μικρό το ποσοστό εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τέλος ο κύριος Τσούμας. Yes, Θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα γενικό σχόλιο ότι όντως βαίνει καλό στο απόθεμα, ενισχύεται διαρκώ, το πιστεύουμε αυτό. Καταρχά, για τελευταίε εκτιμήσει τη επιστημονική Επιτροπή ΣΥΚΑΤ χρησιμοποίησαν τρει διαφορετικέ μεθόδου εκτίμηση για πρώτη φορά που ισχύουν για, όλους, για όλα τα είδη, όνομα τον κόσμο και τα περισσότερα αλληλευτικά είδη που χρησιμοποιεί που αλλιεύει που ενδιαφέρεται, για τα οποία ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν λοιπόν τρεις διαφορετικές μέθοδοι έρευνας τι οποίε εξέθεσα νωρίτερα και θα ήθελα επίση να πω ότι σε συζητήσει με διάφορου αρμόδιους για των αποφάσεων στη συνεδρίαση ΚΑΤ διαπιστώνω ότι εν γέννη επικρατεί η συνένεση πω το 2012 θα γίνει η επόμενη εκτίμηση ε, αποθεμάτων, αποθεμάτων. Και αν επιβεβαιωθεί η αρρωδική τάση των αποθεμάτων θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε και σε αύξηση των ποσοστώσεων αλίευση για το 2013 για τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τη στάση του σε αυτό το θέμα του ερθρού τόνου. Θα ήθελα να πω ότι το επίτευγμα αυτό που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στα αποθέματα, αποθέματα το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, προσπάθειέ του και την πίεση που άσκησαν προ τι ρυθμιστικέ αρχέ ώστε αυτές να κάνουν τη δουλειά του όπως έπρεπε. Όμω από την άλλη μεριά έχουν φτάσει σε ένα σημείο που υπερβάλλουν και είναι και μεροληπτικέ, όπω είπα και στη δική μου ε, παρουσίαση. Η ΚΑΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλες οι αρμόδιες αρχές ε, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά έχουν τα κατάλληλα όργανα, παρατηρούν, παρακολουθούν την κατάσταση, όποιες παραβιάσεις σημειώνονται, τις οποίες άλλωστε υποβάλλουν και στην Επιτροπή Συμμόρφωσης με κυβερνητικές οργανώσεις από πλευρά τους και έτσι λαμβάνεται και η απόφαση από την Επιτροπή Συμμόρφωσης. Άρα ε, θα πρέπει τα σχόλια του κυρίου δίπλα μου να τα λάβετε υπόψη μόνο εφόσον ε, επιβεβαιώνονται και από τις αποφάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Για τις δηλώσεις σχετικές με την Ιαπωνία και τα αποθέματα της Ιαπωνίας, αυτές καλύπτουν δυστυχώ μόνο το ίμιση της αγοράς ε, της Ιαπωνίας για τον τόνο και σε αυτό του δεν είναι αξιόπιστα στοιχεία κατά την άποψή μου. Για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να προσέχετε διότι συνήθως έχετε την τάση να επικεντρώνεται στις ε, θέσεις τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε πελαγικά ψάρια σε μεγάλες ε, ποσότητες, δύο εκατομμύρια τόνους μικρών πελαγικών ψαριών. Μην επικεντρωνόμαστε λοιπόν μόνο στον τόνο, γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε το ρόλο του Θεού. Ευχαριστούμε. Πρέπει να διακόψουμε γιατί ολοκληρώθηκε τη η συνεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση και Εννοείται ότι ο ερυθρός τόνος είναι και το αστέρι των αποθεμάτων ε, στην ΙΚΑΤ, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε την ε, συζήτηση και στο μέλλον. Επόμενο σημείο, έβδομο σημείο, που είναι η έκθεση της που έπρεπε να κάνει η κυρία Λεβάν για τη συνεδρία στη Δισκόφη. Τη ζήτησα και δέχτηκε για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συζήτηση, να αφήσουμε αυτό το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Στα διάφορα ελπίζω να μην έχετε πολλά. Ωραία, ευχαριστώ. Επόμενο θέμα είναι οι αποφάσεις των συντονιστών. Έτσι καλώς σας τις έχουμε μοιράσει. Οπότε νομίζω ότι είναι όλα εντάξει. Δεν βλέπω τίποτα, εγώ δεν βρήκα και κανένα λάθος στις θεσινές μας αποφάσεις. Και τέλος, η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης στο Στρασβούργο στις 4 Απριλίου στις 7 το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για την παρουσία σας και ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Τηρήσαμε την ώρα μας. Καλό σας μεσημέρι.